Uh, uh, uh, Αγαπητοί φίλοι και βουλευτές, ξεκινάει η συνεδρίασή μας. Ησυχία παρακαλώ, για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ. Σας καλωσορίζω όλους. Κάποιο πρόβλημα υπάρχει εδώ διαλύονται καρέκλες. Ωραία. Καλώς ήρθατε. Όλοι οι εκπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων στην συνεδρίαση αυτή την διακοινοβουλευτική που οργανώνει η Επιτροπή Απασχόλησης και βεβαίως καλωσορίζω και τα τακτικά μέλη της Επιτροπής μας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνεδρίασή μας χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο αφορά την, ε, τους δείκτες ε, κοινωνικών θεμάτων και απασχόλησης ε, στην διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών και ειδικά η ανεργία των νέων. Και το δεύτερο μέρος αφορά τον αντίκτυπο του σχεδίου επενδύσεων της Κομισιόν στην απασχόληση. Εάν θέλετε να λάβετε μέρος στην συζήτηση, θα χρησιμοποιήσετε το κίτρινο αυτό φύλλο για τους κοινωνικούς δείκτες και το πράσινο φύλλο αν θέλετε να λάβετε μέρος στη συζήτηση για το επενδυτικό ταμείο. θα προσπαθήσουμε να ακούσουμε διάφορους ομιλητές και έχουμε καθυστερήσει λίγο οπότε η πρότασή μου είναι να ξεκινήσουμε αμέσως τώρα θα πω λίγα λόγια για να ξεκινήσουμε το πρώτο μέρος Πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε την ε, κοινωνική διάσταση όσο και τις μακροοικονομικές πολιτικές. Και είναι φυσικό αυτό βεβαίως για εμάς που είμαστε μέλη της ε, Επιτροπής. Στη χώρα μου, τη Σουηδία, λέμε πως ε, πρέπει να ξέρει η αριστερά μας τι πει η δεξιά μας. Μια τέτοια παροιμία υπάρχει παντού σε όλες τις χώρες φαντάζομαι για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Δεν μπορεί ως βουλευτές ε, να μιλάμε για περισσότερη δικαιοσύνη στην εσωτερική αγορά ενώ από την άλλη να προωθούμε προτάσεις ε, που διευκολύνουν το κοινωνικό ντάμπινγκ στην αγορά εργασίας την φοροδιαφυγή, τον ε, αθέμητο ανταγωνισμό. Μιλάμε από τη μία για την αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης χωρίς από την άλλη να υποβάλουμε προτάσεις έτσι ώστε ο κόσμος να μπορεί να δουλεύει όντως περισσότερο. Προωθούμε, ναι, τις δεξιότητες, επενδύουμε στην εκπαίδευση, ωραία και καλά αυτά, αλλά δεν θα χρησιμεύσουν σε τίποτα εάν δεν επενδύσουμε και στη ζήτηση ταυτόχρονα. Οι αιτίε ε, της ανεργίας των νέων ε, δεν ε, μπορούν να θεωρηθούν μόνο ότι είναι ζήτημα διαφορετικών δεξιοτήτων. Δεν υπάρχουν νέες θέσεις εργασίας από τις οποίες να μπορεί να ζήσει κανείς, όχι μόνο να επιβιώσει και επισφαλείς θέσεις εργασίας. Αυτές δεν φτάνουν δεν μπορούμε να απορριθμίζουμε το εργατικό δίκαιο ειδικά όσον αφορά την ασφάλεια και την υγιεινή συνεργασία για ευελιξία στην αγορά. Αυτό δεν είναι καλύτερη ανάπτυξη. Δημιουργούμε μόνο περισσότερες επισφαλείς θέσεις εργασίας και ο κόσμος μένει σε τέτοιες δουλειές και σε συμβόλαια δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε με χαμηλότερους μισθούς από άλλα μέρη του κόσμου ή με χαμηλότερη ποιότητα ή στις συνθήκες εργασίας. Δεν ανταγωνιζόμαστε την Κίνα, την Ινδία. Για τους νέους, τι σημαίνει αυτό, δεν ξεκινάνε τη ζωή τους. Αν δεν έχουν σταθερή εργασία, δεν μπορούν να νοικιάσουν ένα σπίτι, ούτε τηλέφωνο, το συμβόλαιο τηλεφώνου δεν μπορούν να έχουν, δεν μπορούν να φύγουν από το σπίτι τους και έτσι μετά μειώνεται η κινητικότητα στην αγορά εργασίας και αυξάνεται ο κατακαιρματισμός της κοινωνίας. Για να υπάρχει λοιπόν αηφόρος ανάπτυξη πρέπει να μειώσουμε την ανισότητα. Και αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό για εμάς ε, στις Επιτροπές ε, Απασχόλησης και Κοινωνικών Θεμάτων ε, και στο εθνικό και στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Σήμερα κάποιες χώρες βλέπουν μεγάλα κένα στην κοινωνία που δεν είχαν ξαναδεί από το 1920. Θα έχετε όλοι ακούσει την τελευταία έκθεση της Oxfam που διαπίστωσε πως ο πλούτος του 1% του πλανήτη θα ξεπεράσει το πλούτο του 99% του χρόνου. Πραγματικά πρέπει να το δούμε αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο μας λέει πως ε, αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι συνεργασία και να δούμε συνολικά το θέμα της απασχόλησης. Κανένας νέος δεν θα πρέπει να ξεκινάει τη ζωή του στην ανεργία. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να συντονιστούν και οι ε, δράσεις μας στην αγορά εργασίας και στην οικονομία και ακριβώς αυτό θα κάνουμε τώρα. Όχι μόνο λοιπόν η πτυχή της οικονομίας αλλά ένα κοινωνικό πρόγραμμα Αφού τα είπαμε αυτά λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Μαρία Ντεμαράντζελο Μαρτίνες, εκπρόσωπο της ε, Επιτροπής Δημοσίων Οικονομικών και Δημόσιας Διοίκησης της Ισπανικής Γερουσίας. Ε, μπορείτε να μιλήσετε ισπανικά. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Σά ευχαριστώ που δίνετε την ευκαιρία ούτως ώστε να συμμετάσχω σε αυτόν τον προβληματισμό μέσω τη ισπανική ε, εμπειρία, ιδίω όσον αφορά την απασχόληση. Όπω ήδη γνωρίζετε, η ανεργία είναι η πρώτη μέρημνα τώρα των Ισπανών. Αυτό είναι ευνόητο γιατί εδώ και τρία χρόνια είναι η χώρα που έχουν χαθεί περισσότερε θέσει εργασία στην Ευρώπη. Και αυτά τα τρία χρόνια έχουμε ένα δίκτυο για δημιουργία θέση απασχόληση και είναι η πρώτη μα προτεραιότητα για την κυβέρνηση. Οπότε κατά αυτή την ε, τριετία αυτό το οποίο κάναμε είναι να ξεκινήσουμε κάποιες διαδικασίες όσον αφορά τα, τα δημοσιονομικά μας, όσον ε, αφορά την εξυγίανση του, της οικονομίας μας, αλλά επίσης έχουμε ξεκινήσει και πάρα πολλές μεταρρυθμίσεις για ανταγωνιστικότητα. Και αυτό γίνεται με, ε, γύρω από έναν άξονα που είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και διαπιστώθηκε ότι αυτή την τριετία ε, η κρίση σιγά σιγά έσβησε μέσω αυτών των μετρών των αυτών των μέτρων αλλά και με των προσπαθειών της ε, κοινωνίας μας και με αυτή την ε, αποτελεσματικότητα προσπαθούμε να επιταχύνουμε ε, την αύξηση των ρυθμών ανάπτυξης αλλά και την απασχόληση. Οπότε τώρα είμαστε σε θετικά νούμερα και αυτό δείχνει ότι υπάρχει σταθερά μια αναθρέμα της οικονομίας. Πέρσι το 2014 έπεσαν οι ανέργειες του κάτω των 250.000 και αυτοί οι οποίοι είναι γραμμένοι ε, αυξήθηκαν στους 117.000 όσοι είναι γραμμένοι στα γεωνικής πρόνοιας και επίσης ε, είπαμε ότι έχουμε άλλα ε, από τα 3 εκατομμύρια που ήταν τότε γραμμένοι για επίδομα εργασίας ε, τώρα βγήκαν από το επίδομα ενεργείας περίπου τις 600.000 οπότε βλέπουμε ότι με αυτή την αναθέρωμα της οικονομίας έχουμε τώρα και περισσότερη απασχόληση. Και ποτέ δεν έγινε αυτό τόσο γρήγορα, τόσο άμεσα να δημιουργούν τέτοιε θέσει εργασία και τόσε θέσει εργασία. Και είδαμε το ότι είχαμε αυτή την, την τάση ε, παρά την ανάπτυξη που τρέχει κάτω από 1% και είναι πάρα πολύ ευάλωτη. Αλλά όμως τώρα ε, έχουμε και τις μεταρρυθμίσεις και κυρίως στην αγορά εργασίας. Οπότε όχι μόνο καταφέραμε να ε, έχουμε προηγουμένως μια απόλυτη εργασίας αλλά τώρα έχουμε την ευελιξία που χρειάζεται για την αγορά εργασίας. Η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, ιδίω για τους νέους, ήταν από την αρχή στο επίκεντρο των πολιτικών της κυβέρνησης και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Και έχουμε επομένως ε, έπρεπε να κάνουμε κάτι για την απασχολησιμότητα, για αυτούς που φεύγαν από το σχολείο, ε, τις ευάλωτες θέσεις εργασίας και όλα αυτά ήταν ε, πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Οπότε γι' αυτό και φτάσαμε στους 800.000 περίπου νέου, οι οποίοι ούτε δούλευαν ούτε παίρνουν από κάποια κατάρτιση. Κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ ε, κακό για την αγορά εργασία και βέβαια αυτό ήταν και κίνδυνος αυτοί να βρεθούν σε κοινωνικό αποκλεισμό. Γι' αυτό βρήκαμε κάποια ε, άμεσα μέτρα που ξεκίνησαμε το Φεβρουάριο του 2013 και φτάσαμε στα 100 διαφορετικά μέτρα ούτως ώστε να ε, δώσουμε όθηση στην απασχόληση στην αυτοαπασχόληση αλλά και σε σύναψη θέσεων, ε, συμβάσεων ε, εργασίας αορίστου χρόνου. Και φτάσαμε τώρα στους 400.000 νέους οι οποίοι καλύφθηκαν και ωφελήθηκαν από αυτή την ε, ευκαιρία, από αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Και σήμερα έχουμε 20% συμβάσεων εργασίας τέτοιων, ενώ πριν ήταν κάτω από το 20%. Και όσον αφορά τους νέους κάτω από 25 ετών οι συμβάσεις του χρόνου αυξάνονται και φτάνουμε στο ρυθμό του 25%. Περισσότερες συμβάσεις εργασίας, πρακτικές και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Επίσης, θετικό ήταν το ότι έχουμε αυτό το σύστημα εγγύησης για την νεολαία, κάτι το οποίο δίνει κίνητρα ακριβώς όπως και η στρατηγική που εφαρμόστηκε γενικότερα στην Ισπανία. Χρειάζεται επομένως να στρατευτούν όλοι, αλλά επίσης χρειάζεται να είμαστε αποτελεσματικοί, αποφασιστικοί, όλα τα κράτη, αλλά βέβαια και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και στηρίζεται η ανασυγκρότηση της οικονομίας και στις εθνικές προσπάθειες αλλά και σε πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε κάποιους πόρους για κάποιες πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων. Οπότε και εμείς θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ θετικό αυτό το οποίο θεσπίστηκε, δηλαδή το σύστημα εγγύησης για την νεολαία στη χώρα μας. Τώρα το 2015 θεωρούμε ότι έχουμε προοπτικές καλές, γιατί περάσαμε τη μεγαλύτερη φουρτούνα, αλλά δεν ε, κατεβάσαμε τον πύχη για την κοινωνική πρόνοια. Πάντοτε βρισκόμαστε στα, στα επίπεδα 2010-2011. Το 2015, επομένως, οι πιο ευάλωτοι συνεχίζουν να βρίσκονται στο επίκεντρο των πολιτικών της κυβέρνησης. Δύο παραδείγματα για αυτό το μήνα. Πρώτα-πρώτα, μισονομική πολιτική και φορολογική πολιτική. Είχαμε μία μεταρρύθμιση και μεταξύ 2015-2016 θα μας αποδώσει 9 δις. Αυτά θα πάνε στους επιχειρηματίες και τους εργαζομένους και τις οικογένειές τους με αυτή τη μεταρρύθμιση στόχος είναι να δούμε το πώς αυτά τα μακροοικονομικά μέτρα θα οδηγήσουν σε ευημερία όλων. Μια μεταρρύθμιση που θα είναι πάρα πολύ ισχυρό εργαλείο τόνωσης της οικονομίας. Μια μεταρρύθμιση που περιέχει σημαντικά στοιχεία κοινωνικής πρόνοιας για πολλές οικογένειες, για οικογένειες που ε, έχουν στην οικογένειά τους ε, ιδίως κάποιους ε, ανάπηρους. Οπότε και έτσι βλέπετε ότι είμαστε αποφασισμένοι κανείς να μην εξαιρεθεί από αυτή την αναθέρμα της οικονομίας. Αυτό επίσης δείχνει το πόσο είναι δυνατόν η δημοσιονομική πολιτική να δώσει μειώσει στην ανάπτυξη αλλά και στην κοινωνική συνοχή. Δεύτερο παράδειγμα, έχουμε ένα στρατηγικό πρόγραμμα για ενεργοποίηση της απασχόλησης. Αυτό θα στοχεύσει στους άνεργους μακράς διαρκείας. Μιλούμε για το 60% και εγκρίθηκε στις 15 πρώτου ένα τέτοιο πρόγραμμα για εκείνους από αυτούς που είναι οικογενειάρχες και που εξύντλησαν τα μέτρα προστασίας και άρα έχουν μεγάλη δυσκολία να ενταχθούν στην εργασία. Τώρα θα μπορέσουν να μπουν μέσω ε, ειδικά στοχευμένων, προσωπικά στοχευμένων ε, ε, ε, μέτρων και θα φτάσουμε σε μια ε, υποστήριξη ενίσχυση 426 ευρώ ανά μήνα ανά σύμβαση. Είπαμε λοιπόν, να στηρίξουμε επομένω την πολιτική της πρόνοιας και η απασχόληση άρα είναι η πρώτη προτεραιότητα ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας ξέρουμε όμως τι πρέπει να γίνει λένε ότι το, ο σωστό τρόπο, η, η, σωστή ρότα είναι αυτή που σε οδηγεί στο λιμάνι θες να φτάσει. Αυτό θέλουμε να κάνουμε κι εμεί. Και άρα εμεί θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε για την αναθέρμανση τη οικονομία, ώστε να συνεχιστούν αυτά τα μέτρα. Και βέβαια θα πρέπει να υπάρξει κάποια σταθερότητα που είναι το κλειδί για ε, την αναθέρμανση τη οικονομία και είναι και το κλειδί για να πετύχει κανεί κοινωνική ευημερία. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα δώσουμε το λόγο για δύο λεπτά σε θέλω να μιλήσουν. Κάτριν Σόμπορ, αρχικά από το Ουγγρικό Κοινοβούλιο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι. Εγώ είμαι μέλος ε, της Επιτροπής ε, Ευρωπαϊκών Θεμάτων. Υιοθετήσαμε το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο, είχαμε τακτικά συνεδριάσεις και έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση στην ε, Ευρωπαϊκή Ατζέντα 2020. Θέλουμε να προωθήσουμε την ανάπτυξη και να μειώσουμε την ανεργία. Θεωρούμε πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Άλλα θέματα που μας απασχολούν είναι το σχέδιο επενδύσεων που επικεντρώνεται στη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και βεβαίω οι μικρομεσαίε επιχειρήσει είναι πολύ σημαντικό κομμάτι τη ουγγρική οικονομία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Στην πολιτική συνοχή είναι σημαντικό οι πόροι να μην δαπανούνται αλλού για άλλα έργα από αυτά που είχαν προβλεφθεί αρχικά. Τα έργα αυτά τα που υποτίθεται ότι θα λαμβάνουν χρηματοδότηση, θα πρέπει να τη λαμβάνουν τελικά. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να επικεντρωθούμε και στη, και στη γεωγραφική ισορροπία. Ευχαριστώ. Σε ό,τι αφορά την κατανομή τη χρηματοδότηση. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριος Λούμπα Βλαχά. Από τη Σλοβακία. Έχετε δύο λεπτά, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβαση της Προέδρου. Αναφέρθηκε στην επισφάλεια ως ένα από τα πιο σημαντικά προβλήματα. Συμφωνώ και στη Σλοβακία ε, οι ε, ε, εργασιακές συνθήκες για τους υπαλλήλου αντικαθίστανται από τι εργασιακέ συνθήκε για του αυτοαπασχολούμενου. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα γιατί δεν έχουν ούτε επιδόματα ούτε κοινωνική ασφάλιση. Είναι πρόβλημα και για την κοινωνική ασφάλιση γιατί οι εργοδότες θα, μπορούν, θα έπρεπε κανονικά να ε, καταβάλουν ε, τις ε, απαραίτητες χρεώσεις, αλλά δεν το κάνουν επειδή τους λαμβάνουν ως αυτοαπασχολούμενους. Προσπαθούμε να αλλάξουμε τους νόμους και τους ορισμούς, αλλά επιχειρήσεις πάντα βρίσκουν έναν τρόπο ε, να στραφούν στην επισφάλεια. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα κοινό όραμα πλευρά τη Ευρώπη εναντίον αυτών των καταχρήσεων. Υπάρχει όμω και το πρόβλημα του κοινωνικού ντάμπινγκ, όπω είπατε. Στι χώρε όπω η Σλοβακία, συχνά κατηγορούνται από πλουσιότερε χώρε τη Δύση ότι χρησιμοποιούμε αυτό το κοινωνικό ντάμπινγκ. Όμω βλέπουμε ότι όταν προσπαθούμε να το αλλάξουμε αυτό, πολλέ φορέ οι πρέσβει τη Δύση προσπαθούν να μα πιέσουν για να προστατεύσουν τι ε, δυτικέ επιχειρήσει. Εγώ προσωπικά προσπαθώ να το αλλάξω αυτό και βλέπω πολύ συχνά, προς έκπληξή μου, ότι ε, δέχομαι πιέσεις από τις ε, πρεσβείες της Δύσης. Είναι λοιπόν πρόβλημα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Thank you. Ε, ευχαριστώ. Άντρε Χούνκο από το Γερμαν... τη Γερμανική Βουλή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είμαι από τη Γερμανία, από το κόμμα η αριστερά, δηλαδή αντιπολίτευση, όχι συμπολίτευση. Τώρα μιλάμε για αυτό το νέο μέσο που λέγεται πίνακας βαθμολογίας. Αν δούμε συνολικά τα μέσα που υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει μια ανισορροπία. Δηλαδή αφενός έχουμε μέσα δημοσιονομικής πολιτικής όπως το Δημοσιονομικό Σύμφωνο, το εξαπλό, το διπλό, πακέτο, λίγα μέσα συντονισμού και οικονομικής πολιτικής και ελάχιστα κοινωνικής πολιτικής. Οπότε η βαθμολογία αυτή σύχθη για να υπάρξει κάποια ισορροπία, αλλά νομίζω πως δεν επαρκεί ως μέσο όταν ε, καταρτίζονται δείκτες. Ε, εντάξει, κάτι γίνεται, αλλά δεν περιγράφουμε τις αιτίε ε, και δεν υπάρχει ένας αυτοματοποιημένος μηχανισμός για να αλλάξουμε πορεία, όπως γίνεται με τα άλλα μέσα τα οποία αναφέρθηκαν. Αν δούμε τώρα την Νότια Ευρώπη αναφέρθηκε η κατάσταση στην Ισπανία με ανεργία νέων πάνω από 50%. Ελλάδα το ίδιο. και ε, ε, είδαμε τι έγινε μετά τις ανάλογες αντιδράσεις, οι εκλογές στην Ελλάδα, οι διαδηλώσεις στην Ισπανία, την Κυριακή. Πρέπει λοιπόν να ενισχύσουμε στο ευρωπαϊκό επίπεδο τόσο πολύ την κοινωνική διάσταση έτσι ώστε όταν έχουμε προβλήματα να υπάρχει κάποια αντίδραση, όχι απλά να παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον πρώτο Ευρωβουλευτή, τον κύριο Χαριέρ Λόπες από την Ισπανία. Ευχαριστούμε πολύ. Κάποιες παρατηρήσεις για αυτά τα οποία να μας εξηγήσετε για την Ισπανία και για το πώς έχει κατάσταση στη χώρα. Μήπως ζούμε σε άλλη χώρα. Εγώ εκεί που ζω έχουμε 24% ανεργία και 50% ανεργία στους νέους και εκατοντάδες χιλιάδων που αναγκατέστηκαν, αναγκαστήκαν να μεταναστεύσουν σε άλλες χώρες και αυτές οι μεταρρυθμίσεις που είναι τα τελευταία χρόνια, ιδίως στα εργασιακά συνάντησαν την ε, άγρια αντίδραση των συνδικάτων. Πέρσι δε είχαμε κατά μέσο όρο 54% σύγχρονα 54 ημέρες προσλήψεων και σύγχρονα με τα συνδικάτα πήγαμε πίσω 20 χρόνια. Όχι, δεν είμαι εδώ για να επικρίνω εσάς την κυβέρνηση, αλλά ο ρόλος μας είναι να βρίσκουμε λύσεις αλλά οι λύσεις είναι μακριά από αυτόν τον εφησυχασμό. Δεν κάνει αυτό που απαιτεί η κοινωνία, η κυβέρνηση. Υπάρχει ο αυτός ευάλωτος κόσμος και αυτό μας νοιάζει. Έχουμε 400.000 εξώσεις για στεγαστικά δάνεια. Και αυτό έγινε και από τη δική σας κυβέρνηση και από τη δική μας και αυτό εμένα δεν με πειράζει να το πω. Οπότε αυτή η αναθέρμανση οικονομία από πλευρά ΣΑΕΠ όντως έγινε αλλά ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε στο μέλλον μια ανάπτυξη η οποία ανάπτυξη θα ωφελήσει την αγορά της απασχόλησης. Να μην έχουμε πια αυτή την απαράδεκτη απεργία. Να μην λέει δηλαδή το Δουνουτού ότι έχετε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη αλλά από την άλλη μεριά να έχουμε αυτό το 21% της, ε, της ανεργίας. Δεν είπα ότι φταίτε εσείς, ούτε εγώ φταίω για αυτό που είναι στις οικονομίες μας, αλλά φταίμε όλοι μαζί και οι ανισότητες, το χάσμα πλουσίων φτωχών, όσο πάει και μεγαλώνει. Οπότε αυτό υπονομεύει το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο, την δημοκρατία, την ισότητα. Και αυτό είναι και κάτι σαν διαζύγιο μεταξύ πολιτικής και κοινωνίας. Οπότε ας αφήσουμε επομένως τη μικροπολιτική για τις πολιτικές κουβέντες. Ευχαριστώ. Τώρα έχω μόνο ευρωβουλευτές στο κατάλογο μου. Επομένω, παρακαλώ αν θέλετε να πείτε κάτι, να παρουσιάσετε και την οπτική γωνία των Εθνικών Κοινοβουλίων. Παρακαλώ, ζητήστε τον λόγο. Λοιπόν, κυρία Τετσιάνα Μπέγκη έχει το λόγο, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Παρακαλώ, για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Σε συνέχεια, τον όσο είπαν οι δύο τελευταίοι προλαλήσαντες, να σας επισύρω την προσοχή στο θέμα των δικτών. Η Επιτροπή έχει πει ότι πρέπει να προσέξουμε την κοινωνική πτυχή της ωνέ Και επίσης αυτό θα πρέπει να βοηθήσει για να άρουμε αυτή τη μακροοικονομική ανισορροπία. Υπάρχει ανισότητα και υπάρχει και ο κίνδυνος της φτώχειας. Επομένως, αυτά τα κριτήρια και οι δείκτες μας βοηθούν να συνειδητοποιήσουμε πώς έχει σήμερα η κατάσταση σε κάποια χώρα. Όμως, από την άλλη μεριά, για τις επιλογές της κυβέρνηση δεν βοηθάει και τόσο πολύ. Μπορούμε, επομένως, να προβλέψουμε πώς θα πάει η κατάσταση, μπορούμε να κάνουμε κάποιο είδους συμβουλές επιλογής μακροπρόθεσμες, αλλά τώρα δεν έχουμε απλώς αποτύπωση του σημερινού τοπίου. Ε, όμως μπορεί να βοηθήσει να κάνουμε κάποιες προβλέψεις και πιο χρήσιμο θα ήταν να λάβουμε υπόψη άλλους δείκτες, δηλαδή προσβασιμότητα σε ενημέρωση, τις ανισότητες για τις μισθολογίες ανδρών γυναικών, επίσης και τα ποσοστά της φτώχειας μεταξύ των εχόντων εργασία. Άρα αυτά θα πρέπει να λάβει υπόψη για τις κοινωνικέ πολιτικές το κράτος. Και έτσι να μπορούμε να είμαστε πιο αναλυτικοί, πιο συνεπείς και έτσι να δούμε που κατά προτεραιότητα θα παρέμβουμε, ιδίω όσον αφορά την ενεργεία των νέων για το οποίο αναφερθήκαμε. Είπαμε ότι εδώ χρησιμοποιεί η Επιτροπή και άλλου βοηθητικούς δείκτες να λάβουμε υπόψη την πρόσβαση των νέων στην ε, ανώτατη παιδεία ε, σε σχέση με το ποιοι είναι αυτοί που δεν έχουν δουλειά αλλά και δεν έχουν εγγραφεί και σε κάποιο είδους ε, μαθήματα και δηλαδή κατάρτιση εκπαίδευσης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο ισχύει πάρα πολύ για τις νεότερες γενιές και αυτό που θα ήθελα να είναι μια Ευρώπη που να μην κρίνει τα κράτη μόνο σε περίπτωση υπερβολικού ελλείμματος αλλά και σε περίπτωση υπερβολικής ανεργίας ή ανισότητας. Άρα η Ευρώπη να μην είναι μόνο μια οικονομική ένωση ή μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών αλλά να προσβλέπουν στην Ευρώπη σαν έναν χώρο ευημερία και πλήρους απασχόληση. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Σκύβη Κότρα Κόκομα. Um, um, Από την Κύπρο, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Θα ήθελα να σχολιάσω καταρχήν τη δική σας τοποθέτηση για την έκθεση της ε, Oxfam για, την οικονομική, για τις οικονομικές ανισότητες. Πραγματικά, αφού και εσείς την επικαλείστε, νομίζω ότι θα έπρεπε να αποτελέσει ένα εργαλείο για να κατανοήσουμε όλοι ότι οι πολιτικές και τα μέτρα που έχουν μέχρι τώρα ληφθεί δεν έχουν αντιμετωπίσει τα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ε, ο κόσμος και τα κράτη-μέλη ξεχωριστά στην Ευρώπη δεν θα αναφερθώ στα στοιχεία έχετε πει και εσείς αλλά πραγματικά θεωρώ πολύ σημαντικό να αυξάνουν τα κέρδη των δισεκατομμυριούχων και ο κόσμος συνεχίζει και ο κόσμος που ε, πεινά από την άλλη να αυξάνονται τα ποσοστά εκείνων των ανθρώπων. Ακόμα αν θέλετε να αυξάνονται οι δισεκατομμυριούχοι σε βάρος των εκατομμυριούχων. Αυτό είναι αστείο, δεν μας αφορά, όμως είναι μια πτυχή την οποία θα μπορούσαμε έτσι να κατανοήσουμε και να βάλουμε κάτω. Ε, η διαπίστωση από όλες τις, ε, από όλες τις εκθέσεις αξιολόγησης όπως είναι και η επισκόπηση της ανάπτυξης όπως είναι και όλα τα προγράμματα και οι στρατηγικές έχω αναφερθεί προηγουμένως και στην Ολομέλεια ε, οι στρατηγικές, ε, τα εξάπτυχα, τα δίπτυχα και τα άλλα όλα καταλήγουν και διαπιστώνουν ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Άρα θα πρέπει να μας απασχολήσει το έναν πρώτον και κύριο τα θέματα της ανεργίας, με το να προωθούμε πολιτικές ε, επανακατάρτισης, διαβίου μάθησης, δεν βοηθούμε την νεολαία. Απλά αυξάνουμε την επισφάλεια και την ανασφάλεια κυρίως των νέων ή ε, της διακίνησης των εργαζομένων να μεταναστεύουν από τη μια χώρα στην άλλη βλέπουμε ότι στι πλήστε των χωρών κρατών μελών τη ευρωπαϊκή ένωση υπάρχει ένα ποσοστό ανεργία μπορεί να μην είναι ψηλό όπω σε κάποιε χώρε αλλά υπάρχει σε όλε. άρα το μέτρο τη μετανάστευση των εργαζομένων δεν θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Ε, επίση οδηγούνται με τα διάφορα προγράμματα κατάρτιση ε, τα... οι μισθοί προ τα κάτω θα πρέπει να το δούμε. οι εκποιήσει κατοικιών έχουν αναφερθεί προηγουμένω. στην κύπρο έχουμε τι ιδιαιτερότητε μα. δεν είναι τη ώρα να τι αναφέρω. ακόμα και τι κατεχόμενε από την τουρκία περιουσίε οδηγούνται στην εκποίηση για να αντιμετωπίσει ο κάθε άνθρωπος τα οικονομικά του προβλήματα. Θα μείνω ω εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. I'll give... Ευχαριστώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προσωπώντας την Πορτογαλία. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Γνωρίζετε κι εσείς ότι η Πορτογαλία πέρασε μια δύσκολη περίοδο ευθυγράμμισης. Εξετάζουμε σημαντικούς δείκτες που μπορούν να μας δώσουν ε, ελπίδα για το μέλλον. Εφαρμόσαμε πολλές μεταρρυθμίσεις και εργασιακές μεταρρυθμίσεις που μας βοήθησαν να ενισχύσουμε την απασχόληση. Επομένω τα πράγματα στον τομέα της εργασίας είναι καλύτερα στη σχέση με πριν από δύο χρόνια. Όλα αυτά τα συγκρίνουμε με το 2011 όταν ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή. Εξετάσαμε μεγάλη προσοχή τη διαδικασία και υιοθετήσαμε και ένα έκτακτο πρόγραμμα για να συνοδεύσει τις μεταρρυθμίσεις, κάτι που δεν είχαμε προηγουμένως. Βελτιωθήκαμε λοιπόν, βέβαια δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή την προσπάθεια, καταπολεμούμε όμως την νεανική ανεργία. Έχουμε και ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των νέων σε σχέση και με την επιχειρηματικότητα και έτσι ελπίζουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις απασχόλησης και εκεί. Ευχαριστώ. To, ε, Ευχαριστώ. Μέη Σλόβας από τη Λιθουανία. Παρακαλώ. ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή να μιλώνω ποιόν σας σήμερα. Πράγματι και εμείς έχουμε κάνει πολλά, έχουμε πολλές στρατηγικές, έχουμε πετύχει σημαντικά αποτελέσματα. Ωστόσο, ακόμα κινούμαστε με αργούς ρυθμούς και δεν έχουμε φτάσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κύριο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε αρκετούς πόρους. Για παράδειγμα, στη Σουηδία οι δαπάνες είναι πολλαπλάσιες. 10.000, στη Δανία 11.000. Στη Λιθουανία 208. Η μέση σύνταξη είναι περίπου 1.200 ευρώ. Στη Δανία πολύ παραπάνω. Επομένως, γιατί είδους ασφάλεια θέλουμε να επιτύχουμε. Όταν οι πολίτες ψήφιζαν για την προσχώρηση, την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλαμε την, ε, αυτή την πτυχή της συνοχής, το άρθρο 9 της ε, συνθήκης που μιλά για την ε, κοινωνική ασφάλεια των πολιτών. Η κοινωνική διάσταση συνδέεται απευθείας με την κοινωνική ευημερία. Και αυτό είναι υψή τη σημασία. Η κοινωνική προστασία και ο κοινωνικό τομέα εν γέννη είναι εξαιρετικά σημαντική για κάθε χώρα. Είναι θέματα εθνική ασφάλεια. Και η αυξανόμενη ανέχεια, ιδίω σε μικρότερε χώρες και ο κοινωνικό αποκλεισμό περνά μετά και γίνεται πολιτικός αποκλεισμό. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν. Πρέπει να καθορίσουμε τα ελάχιστα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία. Θα πρέπει αυτά τα πρότυπα να είναι υποχρεωτικά. Για παράδειγμα, η συνταξη θα πρέπει να διασφαλίζεται σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για πολλά ζητήματα θα πρέπει να ανάγονται σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης γιατί αυτό είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Ireland, uh, Την Ιρλανδία έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ενδιαφέρουσες οι παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων. Να πω πως είχαμε και εμείς παρόμοιες εμπειρίες στην Ιρλανδία, αλλά το τελευταίο 1,5 χρόνο καταφέραμε να αλλάξουμε την οικονομία μας. Έχουμε μια ανάπτυξη 5%, η ανεργία από το 15% έπεσε στο 10%, αλλά μου έκανε εντύπωση αυτό το οποίο είπατε και μιλάτε για την Ευρώπη στο σύνολό της και το ε, μέλλον της Ευρώπης ότι δεν θα ε, είναι δουλειές χαμηλής ποιότητας και στην Ιρλανδία όπως και αλλού έχουμε πράγματι πρόβλημα με την αμεβαιότητα στην αγορά εργασίας για τους εργαζόμενους ειδικά όσον αφορά αυτά τα συμβόλαια, τα ορομίστια ειδικά καθώς έχουμε και υπουργό με αυτή την αρμοδιότητα. Αλλά υπάρχει ένα ζήτημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική του 2020. Τονίσαμε το θέμα των ε, θέσεων εργασίας χαμηλής ποιότητας και ότι θα πρέπει να υπάρξει ένας στόχος ποιότητας εργασίας για να δούμε βέβαια και το επίπεδο της ανεργίας. Επίσης αναφέρατε, κυρία Πρόεδρε, πως ε, σε σχέση με τους ε, νέους, πράγματι οι νέοι δυσκολεύονται πάρα πολύ στο να πάρουν ένα σπίτι ή να βρουν στέγη γενικώ. Και βεβαίως εδώ πέρα υπάρχει το πρόβλημα μετά ότι θα έχουμε διαμάχη μεταξύ των ε, γενεών και κόσμος ο οποίος δεν έχει μια ασφαλή θέση εργασίας θα έχει πρόβλημα. Αλλά αυτό σημαίνει πως ε, για να δούμε τους νέους που δεν ε, δουλεύουν ή καταρτίζονται θα πρέπει να δούμε τα πράγματα από κάτω προς τα πάνω. Δηλαδή να ξεκινήσουμε με την εκπαίδευση νωρίς στην παιδική ηλικία. Ειδικά για την ανεργία των νέων πρέπει να τονίσουμε την σημασία αυτή της εκπαίδευσης νωρίς στην παιδική ηλικία. Ευχαριστώ Γιούτα Στάινρουκ, μέλος της Επιτροπής μας εδώ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω συμφωνούμε όλοι στο ότι αν θέλουμε να βγει η Ευρώπη από την κρίση και να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην Ευρώπη θα πρέπει να κάνουμε κάτι για αυτό το θέμα και, και στα εθνικά και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να συμφωνήσουμε στο τι πρέπει να γίνει. Ο κόσμος θέλει κοινωνική ασφάλεια, θέλει να καταργήσουμε και να καταπολεμήσουμε το κοινωνικό ντάμπινγκ, δεν θέλει να αποκλείονται άνθρωποι από την αγορά εργασίας. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας ειδικά για νέους, αλλά βιώσιμες, όχι αυτά τα συμβόλαια, τα ορομίστια. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε από κοινού. Και τον Νοέμβριο δημοσιεύτηκε ακριβώς μια σχετική έκθεση του λεγόμενου Alert Mechanism που έδειξε την ανισότητα και Πραγματικά ένα από τα πιο επίγοντα προβλήματα είναι να μπει η απασχόληση και τα κοινωνικά στο ίδιο επίπεδο με την οικονομική πολιτική και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε τις ε, αναλύσεις και να γίνουν δεσμευτικές οι συστάσεις του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Βεβαίως ε, θα πρέπει να έχουμε κάποιους στόχους για την καταπολέμηση της ε, ανεργίας. Ε, κατά την άποψή μου θα πρέπει πράγματι να συζητήσουμε τους νέους ε, δείκτες, αλλά μην ξεκινήσουμε πάλι να λέμε τι δείκτες χρειαζόμαστε. Με τα μέσα που έχουμε ήδη μπορούμε να κάνουμε κάποια ανάλυση. και πραγματικά να χρησιμοποιήσουμε τους δείκτες αυτούς και να αναλύσουμε τα προβλήματα και να υπάρξει κάποια πρόοδος. Έτσι θα γίνει γιατί μόνο πανευρωπαϊκά μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα από κοινού. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Μπόργκ από τη Μάλτα το κοινοβούλιο εκεί. Χωρίς μικρόφωνο κύριε Σπόρκ. Πατήστε το κουμπάκι για να σας ακούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Μαλτέζος είμαι από τη μικρότερη χώρα της Ένωσης αλλά παρά το ότι η χώρα μας είναι μικρή έχουμε ένα ρόλο να παίξουμε θεωρώ έτσι ώστε να βγει η Ευρωπαϊκή Ένωση από τις δυσκολίες που έχει στη Μάλτα. Θεωρούμε πως η εκπαίδευση είναι το καλύτερο μέσο για κοινωνική ένταξη καθώς ε, έτσι δίνονται τα μέσα εκείνα έτσι ώστε οι οικογένειες, οι εργαζόμενοι να είναι ανεξάρτητοι και να μπορούν να ζήσουν. Στη Μάλτα τα τελευταία δέκα χρόνια περάσαμε από μία περίοδο που έπρεπε να αναδιαρθρώσουμε την ε, οικονομία μας και την αγορά εργασίας η οποία βασίζεται στην ε, βιομηχανία. Επασχολείται πάρα πολλοί κόσμος σε βιομηχανίες και πρέπει να περάσουμε και σε κάποιους πιο εξειδικευμένους τομείς, ε, ηλεκτρονικά παιχνίδια, αεροδιαστημικός τομέας, φαρμακευτική βιομηχανία, τομείς που προσθέτουν ε, προστιθέμενη αξία. Αν όμως δεν είχαμε αυτή την εκπαίδευση και την κατάρτιση θα κινδυνεύαμε με κοινωνικό αποκλεισμό γιατί αυτοί οι εργαζόμενοι που είχαν περάσει όλη τους τη ζωή σχεδόν να δουλεύουν σε κάποιους τομείς δεν θα ήταν ανταγωνιστική. Επίσης παρέχουμε βοήθεια στους αυτοαπασχολούμενους και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντική για την κοινωνία μας και την οικονομία μας και προωθούμε και το επιχειρηματικό πνεύμα καθώς θεωρούμε πως έτσι αυξάνεται η δημιουργικότητα, η ανεξαρτησία, η ελευθερία για να μπορεί κανείς να προοδεύσει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μας βοήθησε, το ότι μπήκαμε στην Ευρωζώνη μας βοήθησε και βεβαίως ε, επενδύσαμε περισσότερο στην αγορά εργασίας και στους εργαζόμενους μας, ελπίζω. Η κυβέρνησή μου τα έξι χρόνια που ερχονται μέσω του πακέτου συνοχής να χρησιμοποιήσει καλύτερα αυτά τα κονδύλια για να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε σε μια ανταγωνιστική αγορά. Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση στον πρώτο γύρο από τον κύριο Πάβελ, Ευρωβουλευτή από τη Ρουμανία. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα αρχικά να αναφερθώ ακριβώς το ίδιο θέμα που θίξατε κι εσείς. Δυστυχώς ε, στην Ευρώπη δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε τους ε, μικρούς μισθούς της ε, Ανατολής. Η νομοθεσία μας επιβάλλει σε συγκεκριμένες εργασιακές συνθήκες. Και έτσι επιβάλλονται αυτές οι συγκεκριμένες συνθήκες. Doar le oferim o piață cu forță de muncă mult mai ieftină și για αυτό το λόγο δημιουργούνται σημαντικά πρόβλημα και όχι μόνο επειδή ε, η εργατική δύναμη είναι πολύ φθηνότερη, για παράδειγμα, σε μια χώρα όπως η δική μου, αλλά και επειδή ε, από κάποιες παρεμβάσεις ε, προτάθηκαν διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε εμά και οι μισθοί και οι φόροι είναι χαμηλοί. Τι μας μένει τελικά, τίποτα για να καλυφθεί αυτό το χάσμα μεταξύ δύση ε, και Ανατολής, μας δίνεται η εντύπωση ότι η Ρουμανία και άλλες χώρες ε, της Ανατολής, επειδή ακριβώς έχουν ε, φθηνότερα εργατικά χέρια, αυξάνεται το κέρδος. Όμως θα πρέπει και ο δυτικός τομέας να καταλάβει ότι αν μειωθεί το κέρδος, θα μπορούσε να αποτελέσει στήριξη για κάποιες χώρες, για τους εργαζομένους τους, ούτως ώστε να μην εγκαταλείπουν τις χώρες τους ε, οι εργαζόμενοι. Γιατί και οι ίδιοι οι νέοι προτιμούν να βρουν δουλειά στη χώρα τους. Γιατί βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμα περισσότεροι νέοι άνεργοι που δεν έχουν ε, γραφτεί στον ΑΕΔ για παράδειγμα, μένουν με τους γονείς τους, με τους παππούδες τους και αυτοί θα ήθελαν ακόμα να κάνουν οικογένεια, αλλά δεν μπορούν ούτε να αγοράσουν ένα σπίτι. Νομίζω ότι η εγγύηση για τους νέους είναι ένα πολύ ε, θετικό σχέδιο και μπορούμε να είμαστε περήφανοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όμω είναι ανεπαρκέ. Γι' αυτό θα πρέπει να δώσουμε πόρου για να διασφαλίσουμε την ανεξαρτησία των νέων. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να διευκολύνουν την πρόσβαση των νέων στο δημόσιο τομέα. το δημόσιο θα πρέπει να δίνει θέσεις για τους ε, νέους που τώρα μπαίνουν ε, στον, στην αγορά εργασίας. Α, έχουμε ακόμα μία παρέμβαση. Μάριο Ρούβο, από την Πορτογαλία. Ενάμιση λεπτό έχει τη διάθεσή σας. Ευχαριστώ. Όλοι κατανοούμε ότι η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης θα πρέπει να ενισχυθεί. Και δεν πρέπει μόνο να εξετάζουμε τα στατιστικά στοιχεία ή την ιδεολογία μας, θα πρέπει να δούμε ότι έχει αυξηθεί η ενεργεία, έχει αυξηθεί η επισφάλεια, ότι με τα μέτρα λιτότητας ε, ε, έχει αυξηθεί ο αριθμός των ανέργων και αυξάνεται όλα και περισσότερο. Νομίζω ότι όλοι το βλέπουμε αυτό. Στην Πορτογαλία έχουμε 35% σε συγκεκριμένους δείκτες ε, ιδίω της νανικής ανεργίας και συνεχώς αυξάνεται τους τελευταίους μήνες. Τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη καταφέραμε, ή μάλλον κατάφερε η, Τρόικα να επιβάλλει μέτρα λιτότητας που δεν ε, ούτε μειώσε την ανεργία, ούτε βελτίωσε τις συνθήκες και γι' αυτό θα πρέπει και η Ευρώπη μέσω του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής ε, να είναι σε θέση να εφαρμόσει κοινωνικά μέτρα που σε άλλες χώρες βοήθησαν ε, να προωθηθεί η πραγματική κοινωνική διάσταση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Thank you very Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση. Μόνο με 1,5-2 λεπτά παρεμβάσεων είναι πολύ δύσκολο να έχουμε μια πλήρη εικόνα της κατάστασης σε όλη την Ευρώπη. Θα αφήσουμε τώρα το πρώτο θέμα της ε, συνεδρίας και θα περάσουμε στο δεύτερο θέμα Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Και χρήση των ε, στόχων απασχόληση για την δημιουργία θέσεων απασχόληση. Ο κύριο Έντμαντ Βίλμπολ έχει το λόγο, πρόεδρο ε, τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της ε, Πολωνικής Γερουσίας. Για πέντε λεπτά έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσω στα πολωνικά. Ε, e, Κυρίες και κύριοι, υπό τη σημερινή συγκυρία κάθε πρωτοβουλία που βοηθάει να αποτελματωθεί η οικονομία είναι ιδέα αξιόλογη ότι έχουμε φτάσει στο 25% ανεργία. Βέβαια, έχουμε 10% πτώση οικονομικής δραστηριότητας. Πάντως, παραμένει το 25% για την ενέργεια των νέων, κάτι που είναι πάρα πολύ ψηλό. Τώρα, για να παραπέμψω αυτό που ακούσαμε προηγουμένω, χρειάζεται για την κατάρτιση μια μεταρρύθμιση. Θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον κόσμο. θα πρέπει να πηγαίνει περισσότερο στα πανεπιστήμια. Εμεί στην Πολωνία επικεντρωνόμαστε στι ε, θετικέ πάση θεωρητικέ επιστήμε. Θεωρούμε ότι αυτό είναι καλή ιδέα. Και η κυβέρνηση λέει ότι είναι αξιόλογο αυτό το σχέδιο για το Ταμείο Στατικών Επενδύσεων της Επιτροπής Γιουνκέρ. Αυτές οι επενδύσεις θα είναι κάτι πάρα πολύ θετικό σε αυτή τη φάση. Για να δούμε τώρα ποια είναι τα επιχειρήματα κατά αυτή της ιδέας. Εάν συνεχιστούν τα παλιότερα προγράμματα, αυτό είναι καλή ιδέα, δικαιολογείται ή όχι. Γιατί μπορεί κανείς να σκεφτεί ότι με ένα καινούριο πρόγραμμα θα έχουμε μια καινούργια αρχή και θα υπάρξει διακοπή των παλαιότερων προσπαθειών. Δεν είναι κανείς βέβαιος για την επιτυχία του νέου διαβήματος. Ας ρίξουμε μια ματιά στην στρατηγική της Λισαβόνας. Αυτή υπήρξε για να γίνουν τα πράγματα καλύτερα. Τελικά όμως αυτό δεν ευωδόθηκε. Πάντως αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να υπάρχει πολιτική βούληση. Αλλιώς επιτυχία δεν μπορεί να υπάρξει. Θα πρέπει επίσης να υπάρχει και συνένεση σε Συμβούλιο και Κοινοβούλιο. Ίσως γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταμάτησε κάποια από τα προγράμματα που καταρχήν ε, έτρεχε ή ήθελε να τρέξει. Οπότε να δούμε τώρα αν χρειάζεται με αυτό το πρόγραμμα καινούργια χρηματοδότηση. Πρόκειται για ένα καινούργιο ταμείο, πρόκειται για καινοτομία, εγγυήσεις και δάνεια. είναι πολύ ψηλό και υπεραισιόδοξο το ποσοστό ομόχλευσης. Μιλάμε για 21 δις. Και 294 ιδιωτικά ταμεία το οποίο θα δημιουργηθούν. Και πάμε άρα στο νούμερο των 350 δις για το μέλλον, για την άμεση φάση. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι αμφίβολο και υπεραισιόδοξο. Και πρόκειται για πρόγραμμα υψηλού κινδύνου. γιατί το ιδιωτικό κεφάλαιο πάντοτε διστάζει πριν προσχωρήσει σε τέτοια διαβήματα. Είχαμε επίσης και την ιδέα την πρώτη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα ομόλογα του 2012. Ο δε 15 είναι επίσης υπεραισιόδοξο. Θα πρέπει το Ταμείο βεβαίως να πρικοδοτηθεί. Βεβαίω και θεωρούμε ότι είναι αναγκαίο αυτό το Ταμείο, αλλά θα πρέπει να διέπεται από υγιείς κανόνες. χρειαζόμαστε να είμαστε πάρα πολύ συγκεκριμένοι στο πώς θα λειτουργήσει το Ταμείο. τα κράτη-μέλη πρέπει να βοηθήσουν. Πρέπει να βοηθήσουν οικονομικά. Τώρα κάτι άλλο. Εάν επικεντρώσουμε την προσοχή μας σε τέτοιες στρατηγικές επενδύσεις ευρωπαϊκές, θα πρέπει να δούμε ποιος ήταν ο ρόλος των ΜΜΕ. Γιατί οι ΜΜΕ δημιουργούν θέσεις απασχόλησης. Και αυτές είναι οι ατμομηχανοί της οικονομίας. Επίσης έχουμε τα ενεργειακά δίκτυα, έχουμε τις μεταφορές, την ε, καινοτομία. το ευρωζωνικό ίντερνετ που είναι όλα αυτά πολύ σημαντικά. Αλλά θα αποδώσουν μακροπρόθεσμα, άρα χρειάζεται υπομονή για να δούμε τους καρπούς αυτών των ε, προσπαθειών. Σας ευχαριστούμε που ακούσατε. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Και τώρα δώσουμε τον λόγο στον κύριο Ντομινικάνιγκαν, ο οποίος ε, είναι Πρόεδρος της Επιτροπής Ευρωπαϊκών του Ιρλανδικού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ. Η ανεργία των νέων είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε. Είπαμε για 24 εκατομμύρια ανέργους σήμερα και πέντε από αυτούς κάτω από τα 25. Όλοι ανησυχούμε ότι θα υπάρξει στασιμότητα στην οικονομία αν δεν έχουμε ανάπτυξη και επενδύσεις. Οπότε είναι πολύ αξιόλογη η πρόταση η Juncker και πάρα ευτυχώς που διατυπώθηκε τόσο γρήγορα με το πανέλαβε τις, ε, τα καθηκοντά του. Όμως θα γίνει με την περιφέρεια της ε, Ευρωζώνης, εκεί που υπάρχει κατά τους ε, επενδυτές μεγαλύτερο ρίσκο. Δεν μιλώ για τις χώρες που επλήγησαν από την κρίση. Το 315-340 θα πάνε σε μακρόπνες επενδύσεις και 75 εκατομμύρια πρόκειται να πάνε σε κάποιες επενδύσεις ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Είναι πάρα πολύ θετικά τα όσα είπε ο ΙΗ συνάδελφο από την ε, Μάλτα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη θέση απασχόληση. είναι πρόβλημα για αυτές. Το είδαμε στην ε, ε, Ιρλανδία ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμπόδιο το τι θα γίνει με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για αυτές τις επενδύσεις. Πάντω, γενικά για όλο αυτό το πακέτο ανησυχούμε. Μιλούμε για 2.000 διαφορετικά, προτάσει. Έχουν υποβληθεί που φτάνουν ε, το 1,5-3, δηλαδή πολύ παραπάνω από την πρικοδότηση. Και είδατε προηγουμένως σε, σε άλλη συνάντηση ότι είπαν ε, οι συναδελφοί σα υπεργών Μπερές και κάποιο άλλο όσον αφορά το ότι υπάρχει πρόβλημα με του ε, επενδυτέ στην Ευρώπη και στην Κίνα. Θα πρέπει να κινηθούμε γρήγορα, θα πρέπει να βρούμε κάποιε λύσει στην κρίση. Αυτό όμω θα απαιτήσει χρόνο για να υλοποιηθεί και τα επενδυτικά ταμεία δεν θα τα έχουμε ή τα χρήματα χρήματο μέχρι το φθινόπωρο, άρα θα πρέπει να υπάρχουν οι δομέ και ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Ξέρουμε ότι από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα προέρχονται τα λεφτά και όπως ξέρετε δεν του αρέσει το ρίσκο και όπως είπε και ο Έντμουντ το πρόβλημα είναι αυτό το 15 προ 1 που είναι η αναλογία τη μόχλευση. Οπότε θα πρέπει να δούμε με προσοχή το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε αυτή τη μόχλευση τώρα οι δαπάνες θα καταμειθούν πολλά χρόνια όσον αφορά κάποια δάνεια για στατικές επενδύσεις συμφωνείτε το αυτό είναι σωστό αλλά θα πρέπει να υπάρχει εξισορρόπηση μεταξύ αυτών των επενδύσεων με το ότι χρειάζεται να δημιουργηθούν τώρα θέσει απασχόληση, ιδίω για του νέου. Είδατε τι είπε ο κ. Λόπε Φερνάντε από την Ισπανία, που είπε για το τι επιπτώσει έχει η ανεργία των νέων. Δεν μπορούν να περιμένουν 7 χρόνια. Όπω είπε και οι συνάδελφοι από την Ιρλανδία, μιλάμε για μια χαμένη γενιά, εκτός εάν ενεργήσουμε ταχύως. Η κυρία Λούμπα από την Σλοβακία είπε για τα δικαιώματα των εργαζομένων, οπότε θα πρέπει οι θέσεις απασχόλησης να είναι βιώσιμες, ποιοτικέ και αυτό μας, ε, ε, μας ανησυχεί, όπως και αυτά τα μηδενικά, συμβάσει συμβάσεις Και έχουμε το θέμα της διαφοράς των ισοτήτων των δύο φύλων, τα είπαμε αυτά συνάντηση του Σεπτεμβρίου και είπαμε ότι θα πρέπει να έχουμε και κοινωνικού δείκτε για την στρατηγική του 2020. Άρα και για αυτή την ιδέα να έχουμε τέτοιου δείκτε που να μα βοηθήσουν να βρούμε βιώσιμε θέσει απασχόληση. Το Δεκέμβριο συμφώνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, άρα τώρα να πιεστούν τα κράτη-μέλη να πρεκοδοτήσουν. Είναι μεγάλες χώρες στην Ευρώπη που μπορούν να επενδύσουν, δεν το κάνουν. Άρα θα πρέπει να τις πιέσουμε για να έχουμε απασχόληση. Κάποιες χώρες, όπως και η Ιρλανδία, έχουν περιορισμό λόγω των κανόνων του Δημοσιονομικού Συμφώνου. Άρα οι επενδυτές θα πρέπει να εξαιρούνται από αυτούς τους κανόνες και με χαρά μου είδα ότι σήμερα είπε ο Γιούνκερ ότι οπωσδήποτε δεν είναι δυνατόν να διέπονται αυτούς τους κανόνες ε, οι επενδυτικές προσπάθειες θα κρυθεί τελικά αυτό το πρόγραμμα από το αποτέλεσμα στην απασχόληση. Άρα θεωρούμε θετικό αυτό το πρόγραμμα να έχει πρικοδότηση, να εφαρμοστεί ταχαίως και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν, να βοηθήσουν το Ταμείο. Και η σωστή διαχείριση θα πρέπει να εξασφαλιστεί και έτσι να αποδώσει η ιδέα καρπούς ταχαίως. και να μπορέσουμε να έχουμε τις επενδύσεις όπως προβλέπεται με κάποια μέτρα που να βοηθούν σε βιώσιμες και ποιοτικέ θέσεις απασχόλησης. Thank you. Ε, Ευχαριστώ. Τελευταία παρέμβαση από την κυρία Ντανούτα Γιάσουλου Γιέγκα, μέλος ε, και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αλλά και εισηγήτρια για πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Μετά από τις ε, δύο λεπτομερέστατες αυτές ε, παρεμβάσεις, καλό θα ήταν να αναφερθούμε πιο γενικώ πώς εμείς ε, στο Κοινοβούλιο προετοιμαζόμαστε για την εφαρμογή του κανονισμού. Θα ήθελα επίσης την παρέμβασή μου να επισημάνω για τις θετικές πτυχές της πρότασης Juncker. Εδώ έχουμε να κάνουμε έναν πολύ σημαντικό κανονισμό σε ό,τι αφορά το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρόκειται για ένα έγγραφο που για χιλιάδες Ευρωπαίους αποτελεί πηγή αισιοδοξία για τη βελτίωση του βιωτικού τους επίπεδου. Το έγγραφο αυτό είναι μια ευκαιρία αλλά και ευθύνη που θα πρέπει να υπομισθούμε. Τα όσα προβλέπονται στον κανονισμό είναι να διαμορφώσουμε μια νέα κινητήρια δύναμη ανάπτυξης στην Ευρώπη από την αρχή της κρίσης στην Ευρώπη και εδώ στο Κοινοβούλιο και αλλού τα έχουμε συζητήσει διεξοδικά. Και ελπίζαμε ότι ένα νέο μέσο θα μας δώσει περισσότερη βοήθεια και ελπίδα για το μέλλον. Ήδη σήμερα βλέπουμε ότι δεν καταφέραμε και πολλά σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη, δυστυχώς. Παρά το ειδικό βάρος και τη σημασία του εγγράφου αυτού δεν έχουμε πολύ χρόνο να το επεξεργαστούμε. Ίσως αυτό να είναι καλό γιατί συχνά δεχόμαστε επικρίσεις ότι είμαστε ε, ιδιαίτερα βραδικίνητοι ό,τι αφορά την υιοθέτηση σημαντικών αποφάσεων. Αλλά και εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο δεν έχουμε χρόνο, αλλά και σε άλλα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα δεν υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και να σας υπενθυμίσω όσα έχουν ήδη γίνει και όσα θα γίνουν στο άμεσο μέλλον. Ο πρόεδρο της Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούγκερ, παρουσίασε το σχέδιο επενδύσεών του στα τέλη Ιουλίου του 2014. Το Συμβούλιο θέτησε το σχέδιο το Δεκέμβριο και κάλεσε τους νομοθέτες να ολοκληρώσουν όλο το απαραίτητο έργο μέχρι τα τέλη Μαρτίου. Ταυτόχρονα ο Επιτρόπος Νταμπρόφσκης ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρξει γρήγορα συμβιβασμό με την απαραίτητη στήριξη των κρατών μελών. Οι διαπραγματεύσει ξεκίνησαν στις 19 Ιανουαρίου. Η Επιτροπή μας θα ψηφίσει λογικά την γνωμοδότηση την 1η Απριλίου το αργότερο. Αυτό μας δίνει ε, δύο μήνες για να διαμορφώσουμε μια ισχυρή θέση στην Επιτροπή μας. Αν δεν αλλάξει κάτι, θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι εργασίες επί του εγγράφου έως τα μέσα Μαΐου. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι το Ταμείο θα μπορεί να ξεκινήσει τις λειτουργίες του τον Ιούνιο. Ταχύτατο αριθμός λοιπόν προόδου για μια νομοθετική πράξη. Ο κανονισμός που προτείνει ο κ. Γιούνκερ συμπεριλαμβάνει σωρία θετικών στοιχείων. Το Ταμείο Επενδύσεων βασίζεται σε τρει πυλώνε. Ο πρώτος πυλώνας προσδιορίζει ότι θέλουμε ε, να δώσουμε όθηση σε επιπλέον επενδύσεις για τα επόμενα τρία χρόνια της τάξης των 350 δις ευρώ. Δεύτερος πυλώνας, να έχουμε στοχευμένες πρωτοβουλίες για να διασφαλίσουμε ότι οι πόροι μας ανταποκρίνονται στις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας. Τρίτος πυλώνας, κανονιστική ασφάλεια και προβλεψιμότητα. Θα πρέπει να εξετάσουμε και τον ε, πολλαπλουσιαστικό συντελεστή, εάν περισσότερα κράτη-μέλη συμμετάσχουν στο πρόγραμμα και μιλώ και για ιδιωτικούς επενδυτές και για ε, εθνικές τράπεζες. Οι βασικές έννοιες ε, του Ταμείου μας επιτρέπουν να θεωρήσουμε ότι τα χρήματα αυτά θα δαπανηθούν ορθώς. γιατί βλέπουμε ότι ε, οι πόροι που δαπανώνται για μακροπρόθεσμους στόχους δεν αποδίδουν ε, τα επιθυμητά αποτελέσματα. Οι πόροι που δαπανώνται για την ενέργεια, για τις υποδομές και άλλα project ε, είναι χρήματα που δαπανώνται για την πραγματική οικονομία και έτσι είναι πολύ θετικό. Τα πρώτα θα βασίζονται στην αποδοτικότητά του, στην κερδοφορία του, στην ευρωπαϊκή προσταθεμένη αξία και συμμόρφωση με του ευρωπαϊκού ε, στόχου πολιτική. Τέτοιε επενδύσει έχουν ω στόχο τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόληση. Όμω, η στήριξη δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο σε διασυνοριακά έργα. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μέχρι και 2,5 εκατομμύρια θέσεων απασχόλησης. Οι Ευρωπαίοι και τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα ξέρουμε ότι έχουν ε, περίπου 200 ε, δις ε, σε αποταμιεύσεις σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Έχουμε πολλά χρήματα που δεν δαπανώνται για την χρηματοδότηση πολύ σημαντικών έργων. Και αυτό επειδή ακόμα αντιμετωπίζουμε μια κρίση αξιοπιστίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το νέο Ταμείο Επενδύσεων έχει ως στόχο να μας βγάλει από αυτό το τέλμα στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο μια ελπίδα αυτή, είναι μια πραγματική προσδοκία από πλευρά των επενδυτών. Τώρα, η συμβολή των κρατών μελών στο Ταμείο δεν θα πρέπει να επιβαρύνει περαιτέρω ε, τα ελλείμματα. Κάτι το οποίο θα μας απασχολήσει περαιτέρω. Εμείς εδώ στο Κοινοβούλιο ακόμα έχουμε κάποιες αμφιβολίες για το κατά πόσο ο υποτιθέμενος πολλαπλασιαστής είναι εφικτό να επιτευχθεί. Γιατί έχουμε το πολύ βασικό ρόλο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία σε ό,τι αφορά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Ακριβώς, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κύριοι δικαιούχοι στήριξη από το Ταμείο. Αλλά τίθεται το ζήτημα κατά πόσο τέτοιε μικρομεσαίε επιχειρήσει θα καταφέρουν να δημιουργήσουν τον απαιτούμενο αριθμό και τον απαιτούμενο πολλαπλασιαστή. Η Επιτροπή Επενδύσεων στο πλαίσιο του Ταμείου θα είναι υπεύθυνη για την επιλογή των έργων. Ελπίζουμε να μην κρίνει με πολιτικά κριτήρια, αλλά με βάση τα πλέον αποθετικά έργα. Άλλο πιθανό πρόβλημα είναι η σύνθεση ε, του Διοικητικού Συμβουλίου, του οργάνου που ε, θα αναλάβει την διοίκηση του Ταμείου. Πρέπει να δούμε ποια κρατημέλη θα αναλάβουν τι θέσει αυτές, γιατί η συμβολή του θα είναι και μεγαλύτερη. Λογικό είναι αυτό, αλλά πρέπει να το εξετάσουμε. Θα πρέπει λοιπόν να χρηματοδοτούνται τα πλέον αποδοτικά και προσοδοφόρα έργα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως ακόμα δεν έχουμε συγκεκριμένα κριτήρια για την επιλογή των έργων. Τέτοιε πληροφορίε θα πρέπει να είναι ήδη διαθέσιμε ούτω ώστε πιθανοί επενδυτές να μπορούν να μελετήσουν ε, κατά πόσο έχουν συμφέρον σε αυτό το ταμείο και τα project. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ενδιαφέροντα αυτά που μα είπατε. Τώρα περνάμε στα δίλεπτα. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Γιάκο Μπλούντ από την Δανία και τη Βουλή της Δανίας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εκπροσωπώ του σοσιαλδημοκράτες ε, στη Δανία. Εμείς θεωρούμε πως υπάρχουν ε, αρκετές ε, καλές δυνατότητες για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων. Να δούμε τώρα τι έργα θα εγκριθούν. Ελπίζω να είναι κάποια έργα τα οποία θα αυξήσουν τη ροή της ενέργειας στην Ευρώπη, καλύτερη κατανομή της ενέργειας με τον καλύτερο τρόπο. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για εμένα όταν μιλάμε για τέτοιες επενδύσεις ε, διεθνείς ε, διασυνοριακές ε, είναι ότι θα πρέπει να σεβόμαστε τις συνθήκες ε, της αγοράς εργασίας ε, στα κράτη-μέλη για να μην υπάρχει κοινωνικό ντάμπινγκ. Και ελπίζω πραγματικά να δώσουμε βάρος σε αυτό το κριτήριο. Δηλαδή να εκπαιδευτούν όσοι θα λάβουν μέρος, να αυξηθεί η εκπαίδευση και η κατάρτιση των νέων ε, αλλά και των εργαζομένων γενικώ ε, και να διασφαλίσουμε πως πραγματικά θα εκμεταλλευτούμε πλήρως αυτά τα έργα ενέργεια και υποδομές της ενέργειας. Λοιπόν, νομίζω πως είναι το μις ε, στους οποίους θα επωφεληθούμε και πραγματικά αναμένω εδώ τι θα γίνει. Ευχαριστώ. Θα δώσω τον λόγο στον Σασκι Ουρίνσκας από την Λιθουανία και την Βουλή της Λιθουανίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ένα σύντομο σχόλιο για την ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων και την νεολαία. Είναι αυταξία η ελεύθερη διακίνηση των εργαζομένων. Είναι κάτι το θετικό για όλους. Η χώρα μου, η Λιθουανία, βλέπει πραγματική έξοδο των νέων και ο λόγος είναι η απαράδεκτη οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην ε, χώρα μας. Είναι πολίτες μας, ε, έχουμε επενδύσει, αυτούς τους εκπαιδεύουμε και φεύγουν από τη χώρα γιατί έχουμε μία Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Το τεράστιο χάσμα μεταξύ πλουσίων χωρών, αφενός όπου οι νέοι αυτοί από τις χώρες μας αυξάνουν το ΑΕΠ αυτών των χωρών και όχι της δικής μου χώρας. Είμαστε χαμηλά στον δίκτυ της ε, φτώχειας, αλλά ψηλά στον δίκτυ των αυτοκτονιών. Αυτοί οι νέοι λοιπόν αυξάνουν το ΑΕΠ των ξένων χωρών και κατηγορούνται για τα οικονομικά προβλήματα στις χώρες αυτές, π.χ. στο Ηνωμένο Βασίλειο, πραγματικά είναι εξευτελιστική η κατάσταση. Και η αποδημία τους μειώνει τις οικονομικές μας δυνατότητες, αυξάνει τα δημογραφικά μας προβλήματα και αυξάνει τα προβλήματα των ηλικιωμένων. Προκύπτει λοιπόν ένα ερώτημα. όπως πρέπει να δούμε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή να δούμε τι γίνεται με την έξοδο των εκπαιδευμένων νέων μας, των μορφωμένων νέων μας στις πλούσιες χώρες. Ίσως χρειάζεται μια υποχρεωτική συνοχή, ένας μηχανισμός συνοχής που θα καλύπτει όλη την Ένωση ανεξαρτήτως του εάν ε, μια χώρα είναι φτωχή ή πλούσια. Αυτό θα πρέπει να είναι το κριτήριο. Ευχαριστώ Σίλβια Σύνφα από την Βουλή της Λετωνίας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε αλλαγές ε, στην Ευρώπη, η κοινωνική διάσταση πλέον της ε, ΟΝΕ είναι κάτι το απολύτως αναγκαίο για να μην χαθεί η ορμή και η πολιτική βούληση για να γίνουν αυτές οι βελτιώσεις. Ε, πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία των οικονομικών και κοινωνικών πτυχών με τις μακροοικονομικές πτυχές. Αυτό είναι ιδιαίτερος επίκαιρο. Πρέπει να επιτύχουμε μια συμφωνία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εφαρμόσουμε ένα πακέτο ανάπτυξης και απασχόλησης στο οποίο ελπίζουν πάρα πολύ για να υπάρχει λοιπόν βιώσιμη ανάπτυξη θα πρέπει να έχουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα επενδύσεων και να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα αυτά σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Θα πρέπει λοιπόν οι επενδύσεις ε, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας υψηλής ε, ποιότητας. Κατά την άποψή μου θα πρέπει να δημιουργήσουμε ευνοϊκές συνθήκες για τις εταιρείες και να τις επιτρέψουμε να παίξουν το ρόλο που μπορούν για να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Για να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους πρέπει να βελτιωθεί η χρήση των μέσων κοινωνικού διαλόγου και να βρούμε κάποιες λύσεις για το πώς ε, θα συνεργαστούμε με τους ε, κοινωνικούς εταίρους ε, στην ΟΝΕ και να αποκτήσει, όπως είπα, μια κοινωνική διάσταση. Τείτε επίσης καλύτερη εμπλοκή των εταίρων στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο εθνικό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαρία Χαουροντρίκης από την Πορτογαλία, Ευρωβουλευτής, έχει τον λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι που όλοι ε, οι περισσότεροι συμφωνούν πως χρειαζόμαστε αυτό το επενδυτικό σχέδιο για να έχουμε περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας για την Ευρώπη. και ακριβώς θα πρέπει να δώσουμε μέσα για την ευρωπαϊκή στρατηγική, για την ανάπτυξη και τις δουλειές για να λειτουργήσει, γιατί δεν είχαμε μέσα. Θα πρέπει λοιπόν πρώτα απ' όλα στα κριτήρια επιλογής των έργων να έχουμε σαφή κριτήρια για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ποιότητα των θέσεων εργασίας. Και βεβαίως ε, να χρησιμοποιήσουμε τα κριτήρια αυτά για να αξιολογήσουμε το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Δεύτερον, πάρα πολλοί συνάδελφοι εκφράζουν ανησυχίες για τη δυνατότητα μόχλευσης του ταμείου αυτού. Υπάρχει ο κίνδυνος να μην λειτουργήσει το ταμείο και γνωρίζουμε πως μια προϋπόθεση για ισχυρή μόχλευση είναι οι συνεισφορές των κρατών μελών. και ελπίζουμε οι κυβερνήσεις μας πραγματικά να συνεισφέρουν. Αλλά γι' αυτό θα πρέπει να φροντίσουμε όλα τα κράτη-μέλη να μπορούν να ε, επωφεληθούν από αυτό το ταμείο, κάτι το οποίο ακόμα δεν είναι σαφές. Γιατί όταν ένα κράτος μέλος έχει μία διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος, ε, δεν μπορεί να έχει να εξαιρέσει τη συγχρηματοδότηση των έργων από την πειθαρχία του Ταμείου του Συμφώνου Ανάπτυξης. Τέλος, αλλά σημαντικό, είναι σημαντική αυτή η συζήτηση σήμερα γιατί πρέπει να υπάρχει συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκού και Εθνικών Κοινοβουλίων ακριβώς για να λειτουργήσει αυτό το επενδυτικό σχέδιο πρέπει να ξέρετε πως η ομάδα μας ε, για να στηρίξει τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έβαλε ως όρο να έχουμε ένα επενδυτικό σχέδιο. Ευχαριστώ. Πιότρ Ναϊμίσκι έχει τον λόγο, βουλευτής από την Πολωνία. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω πολωνικά. Το επενδυτικό αυτό σχέδιο έχει στόχο την κινητοποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας, οπότε χρειάζεται αύξηση του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Όπως είπε και η κυρία Ουλφσκοκ, πρέπει να ξέρει η ε, δεξιά μας τύπη, η αριστερά μας, η παραγωγικότητα τώρα και το ποσοστό της βιομηχανικής παραγωγής ως ε, ποσοστό του ΑΕΠ ε, εμποδίζεται από την κλιματική μας πολιτική που είναι ένας έξτρα φόρος εάν θέλετε που εμποδίζει την βιομηχανία. Ένα άλλο ζήτημα τώρα. Τα χρήματα για το σχέδιο του Γιούνκερ από ό,τι κατάλαβα θα αφαιρεθούν από υφιστάμενα έργα που ήδη εφαρμόζονται. Στην ε, Πολωνία, παραδείγματο χάρη, ε, θα φύγουν από το Ταμείο Συνοχής. Δεν πρέπει να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Εντάξει, η γενική κατεύθυνση είναι καλή, αλλά θα πρέπει να δούμε και τις ιδιαιτερότητες των ε, κρατών μελών. Και τώρα έχουμε διάφορα σχέδια για την φορολογική εναρμόνιση που δεν λαμβάνουν όμως τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών και θα εμποδίσουν τις επενδύσεις ή την δυνατότητα επενδύσεων και βεβαίως ε, θα πρέπει να ενισχυθούν από το σχέδιο Juncker. Έχουμε χαμηλούς μισθούς στην Πολωνία σε σύγκριση με το πόσο δουλεύει ο κόσμος και του του η εναρμόνιση του βασικού μισθού στο σημείο 21-33 στο ψήφισμα είναι λάθος, δεν θα πρέπει να γίνει. Ευχαριστώ. Γκαμπριέλα Κρέτσου από την Ρουμανία. Έχετε τον λόγο για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για τις μεταρρυθμίσεις αγορές το δικό μου συμπέρασμα είναι το εξή. Η εγχείρηση πέτυχε, άλλο ο πέθανε πέθανε. Here. For me it's not clear. Ε, για μένα ε, όλα αυτά σημαίνουν για δύο λόγους. Γιατί πρώτα πρώτα δεν έχουμε αγορά απασχόληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε 28 αγορές απασχόλησης με 28 διαφορετικά μισθολογικά επίπεδα, συλλογικέ συμβάσει ή αλλού δεν έχουν συλλογικέ συμβάσει κλπ. Εγώ προέρχομαι από μια χώρα όπου ο μέσος μισθός είναι έξι φορές χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μεσόρο. Και το κόστος διαβίωσης 75-80% του ευρωπαϊκού μεσόρου. Οπότε τα πράγματα δεν είναι σαφή γιατί η αγορά απασχόληση δεν είναι μια αγορά. Ξέρετε γιατί. Γιατί η πλήρης απασχόληση δεν είναι αυτός ο σκοπός. Της ε, οικονομίας αγοράς, της κοινωνίας αγοράς. Είναι κάτι το οποίο εξαρτάται από άλλες αγορές. Την εσωτερική αγορά για εμπορεύοντα και υπηρεσίες. Βασικά αυξάνεται η ζήτηση. Πρέπει όμως να ε, αρθούν οι ανισότητες εισοδήματος. Τότε θα έχουμε απασχόληση. Και αυτό που έχει σημασία είναι η ζωή των πολιτών. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δημιουργούν ε, το 80-90% όπως είπαν και όλοι των θέσεων απασχόλησης. Οι μεγάλες επιχειρήσεις όχι. Δεν δημιουργούν πολλές θέσεις απασχόλησης. ή είναι προσανατολισμένο προς τις ΜΜΕ το σχέδιο Γιούνκερ Καθόλου. Φτιάχνουν λοιπόν ε, αγαθά και υπηρεσίες για τον κόσμο, όμως ο κόσμος δεν έχει χρήματα. Και έτσι αυξάνεται το χάσμα και χρειάζονται μεταρρυθμίσεις. Τι θα πει αισιόδοξο, ένας αισιόδοξο ο οποίος όμως είναι ενημερωμένος. Ακόμα και αν επιβληθεί δια της βίας το σχέδιο Γιούγκερ δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα της ε, ανεργίας που έχουμε. Δυστυχώς. Η πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δώσουμε το λόγο στην Λαώρα που είναι μέλος Επιτροπής μας και Ευρωβουλευτής. Ευτυχώς βλέπω ότι και άλλοι σκέφτονται σαν και εμένα γιατί στο παρελθόν ε, έχω βρει ότι μου είναι ξένες, αλλά δυστυχώς μένουμε στον ίδιο κόσμο και οπότε θα πρέπει να δούμε ότι είναι περίπλοκη κατάσταση όσον αφορά αυτό το νέο ταμείο για τις επενδύσεις. Αυτό του Πρόεδρου Γιούνκερ όμως θα πρέπει συνέχεια να λέμε πόσο είναι κρίσιμη η κατάσταση. Κάποιος να μας πει ότι αυτό είναι θεμητό σκοπός, αλλά Αυτέ οι πόροι ήδη έχουν διατεθεί και θα τις πάρουμε από τη μία τσέπη να τις βάλουμε στην άλλη. Οπότε κόβουμε χρήματα από προγράμματα όπως το Horizon και αυτοί οι πόροι θα πάνε σε αυτό το νέο ταμείο. Για πέστε μου, για εξηγήστε μου. Από πού και ως πού. Αυτό είναι λογικό. Κόβουμε δηλαδή από την έρευνα και τα πάμε κάπου αλλού αυτά τα χρήματα. Μιλάμε τώρα για τον ιδιωτικό τομέα ιδιωτικές επενδύσεις. Μα αν είναι υψηλού ρίσκου αυτή η υπόθεση, ποιος ιδιωτικό τομέα θα κάνει τέτοιες κινήσεις. Μέχρι σήμερα κανένας δεν έχει κάνει τέτοιες ε, κινήσεις. Μα πώς. Είναι δυνατόν έτσι με, το, με την παγκέτα του μάγου να βρούμε χρήματα και επενδύσεις. Μιλούμε για συμμετοχή, συμβολή των κρατών μελών. Και εγώ αναρωτιέμαι, αυτά τα έργα τα οποία επελέγησαν έχουν κάποιο σχέση με τις περιφέρειες. Καμία ασφάλεια δεν διαπιστώνω. Από πού και πού να εγκριθούν αυτά τα σχέδια και προγράμματα. Μα ίσως ε, βοηθήσουν να προχωρήσουν κάποιες χώρες. Εντάξει, να έχουμε ελεγγύη. Αλλά... Αλλά... να μην είμαστε γενναιόδοροι μέχρι ε, παράνοιας, οπότε έχουμε διάφορες περιπτώσεις όπου ε, ε, υπάρχουν κάποια κρατημέλη που έχουν κάποιες ανισότητες, κάποιες έχουν κάποιο χάσμα στα δημοσιονομικά τους με αυτό το έλλειμμα σε σχέση με το ΑΕΠ αλλά τελικά όλο αυτό το διάστημα είδατε πόσο δεν απέδωσαν όλα αυτά τα μακρόπουνα σχέδια. Τίποτα δεν είναι για την ανάπτυξη. Εδώ μάλλον για ακόμα μια φορά πάμε σε βατερλό. Ευχαριστώ. Ούρος Πρίτελ από το Σλοβενικό Κοινοβούλιο. Έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ε, ναι, Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, για να παίξουμε επιτέλους έναν προληπτικό ρόλο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ και για την οργάνωση της σημερινή ημέρας. Σε αντίθεση με τους προλαλήσαντες, που ήταν αρκετά απεσιόδοξη όπως και οι συνάδελφοι από την ε, Ρουμανία εγώ είμαι αισιόδοξο ε, για την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας ε, και για την σταθερότητα και την ποιότητά τους και παρόλα αυτά έχω κάποιες επιφυλάξεις ακούσαμε πως υπάρχουν 24 εκατομμύρια άνεργοι αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και τι να σου πω αυτό είναι 12 φορές η Σλοβενία Βεβαίω ε, συχνά έχουμε και ψηλούς στόχους για την ενέργεια, τις υποδομές, έργα με μεγάλο πολλαπλασιαστή και προστιθέμενη αξία αλλά αυτή την στιγμή θα πρέπει να κινητοποιηθούμε αμέσως. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν κατηγορίες δύο, ε, να υπάρχουν πολίτες με συγχωρείτε δύο κατηγοριών. Ή μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Τέλος θα ήθελα να πω το εξής. Είμαι αισιόδοξο και όλοι μαζί από κοινού οι εκπρόσωποι της Κομισιόν του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου των Εθνικών Κοινοβουλίων και Κυβερνήσεων θα καταφέρουμε οπωσδήποτε να βρούμε κάποιες ισορροπημένες λύσεις, να φτιάξουμε δρόμους και σιδηροδρόμους και οπωσδήποτε να διασφαλιστεί η εργασία για όλους νέους και λιγότερο νέους. Σας ευχαριστώ κυρία Τανκεβίτσιούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να καλωσορίσω και εγώ τους συναδέλφους. Είναι καλό που έχουμε αυτή τη δυνατότητα οι ευρωβουλευτές να συζητάμε με τους βουλευτές ε, για το σχέδιο αυτό Γιούγκερ για τις στρατηγικές επενδύσεις. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενοι συνάδελφοι, κυρίως γιατί η Επιτροπή του Μπαρόζο είχε στόχο να κάνει οικονομίες ειδικά στην κοινωνική διάσταση. Είχαμε λοιπόν αυτό το σχέδιο επενδύσεων που συζητούσαμε εδώ στο Κοινοβούλιο και είχαμε συζητήσει το ότι το επενδυτικό αυτό σχέδιο πρέπει να αποδίδει ως επένδυση και να έχουμε βεβαίως ποιοτικέ θέσεις εργασίας. Το είπαν οι συναδελφοί αλλιώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να αναπτυχθεί, δεν θα υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη και δεν θα έχουμε κανένα αποτέλεσμα και οι τομείς που χρειάζονται επενδύσεις είναι αυτοί που ενισχύουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ασφαλειά της, ειδικά δεδομένης της τρέχουσας γεωπολιτικής κατάστασης ενέργεια, μεταφορές, ψηφιακή αγορά, όλα αυτά που αφορούν ε, την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εάν αποκλείσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν θα επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Και τώρα μιλάμε με τους εθνικούς βουλευτές και τονίζω πως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να είναι σε αυτό το επενδυτικό σχέδιο γιατί βεβαίως αποτελούν τις περισσότερες ε, δημιουργούν τις περισσότερες θέσει εργασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο να βρούμε αυτά τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ τα εθνικά κοινοβούλια όμως οι εθνικές επενδύσεις, οι κοινωνικοί εταίροι όλοι πρέπει να δουλέψουν χέρι με χέρι για να επιτύχουμε τα αποτελέσματα. Ευχαριστώ. Enrique Calvet is... Enrique Calvet δεν είναι εδώ, από ό,τι βλέπω. Ευρωβουλευτή επίση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Περίμενα να ε, ακούσω την μετάφραση. Ε, δεν άκουσα το όνομά μου. Σύντομα να σας πω τρεις σκέψεις μου. Από ό,τι φαίνεται όλοι συμφωνούμε ότι το σχέδιο Γιούγκερ είναι ε, καλύτερο από το τίποτα όσο και αν δεν είναι τόσο φιλόδοξο. Για να δούμε τώρα. Από σκοπιά τελείως πρακτική. Δεν ποιες είναι δυσκολίες να δούμε τι γίνεται. Βραχυπρόθεσμα και τι γίνεται μέσω μακροπρόθεσμα. Όλοι συμφωνούμε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες επενδύσεις που μέσω μακροπρόθεσμα να είναι παραγωγικές, να δίνουν οικονομίε οικονομίες κλίμακας, εξωτερικές οικονομίες, να γεννούν ανάπτυξη κλπ. Όμως με βράχη πρόθεσμα το θέμα είναι η ανεργία. Αυτό είναι το ευρωπαϊκό πρόβλημα, όχι εθνικό γιατί μας οδηγεί σε διάλυση της κοινωνίας και γκρεμίζει το όραμά μας για μια ευρωπαϊκή κοινωνία. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη την ώρα της επιλογής, της απόφασης, οπότε εδώ πέρα υπάρχει πρόβλημα ε, περιχαράκωσης ε, αυτού του προγράμματος. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να επιληθεί. Δεν είναι πρόβλημα χωρών. Το θέμα είναι με τι κριτήρια, από ποια σκοπιά θα προχωρήσουμε το πρόγραμμα. Να γίνει αυτό από πλευρά απασχόλησης. Οπότε εγώ προτείνω να έχουμε κάποια υποχρεωτικά κριτήρια σε σχέση με την απασχόληση. Άμεση, έμεση και επομένως να λαμβάνουμε υπόψη την εμπλοκή των ΜΜΕ που θα δημιουργήσουν τις εργασίες. Χωρίς βέβαια να ξεχνάμε ότι και οι ΜΜΕ επίσης είναι στο, στο, να είναι στο βεληνικέστος των αυτών των μεγάλων των επενδύσεων. Τώρα, μια που πιέζει ο χρόνος τελευταίο, με προβληματίζει το ότι συνέχεια μιλάμε για ποιοτικές θέσεις απασχόλησης, για η απασχόληση βιώσιμη κλπ. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά φυσικά και η ευημερία δεν το συζητώ. Αλλά όμως το πρόβλημα της ανεργίας κάπου στην Ευρώπη να μην θεωρείται ότι είναι πρόβλημα αυτών των εργαζομένων. Αυτό που δεν μπορεί να μην έχουν κατάρτιση κλπ. κλπ. Θα πρέπει και αυτούς να τους καλύψουμε με δημιουργία απασχόληση. Ευχαριστώ, Εμίλιαν Πάβελ, από Ευρωκοινοβουλίου. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον ε, τις προτάσεις ε, και από τους συναδέλφους από τη Ρουμανία και από τις γειτονικές χώρες και βλέπω ότι δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στις υποδομές. Βεβαίως, βραχυπρόθεσμα, οι υποδομές θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν ε, να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες που έχουμε στην απασχόληση. Αλλά θα πρέπει η έμφαση παρόλα αυτά να δοθεί στην καινοτομία, στην έρευνα, στο μέλλον και στην προστιθέμενη αξία που μπορεί να μας δώσει το μέλλον. Από κοινού, με την ενέργεια, ε, την πληροφορική, συμφωνώ πάρα πολύ. Αυτά τα έργα έχουμε ανάγκη. Όμως, ως μέλος και αυτής της ε, Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ή μάλλον η δική μας Επιτροπή θα έπρεπε να προσδιορίσει συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα υποβάλει ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κριτήρια επιλεξιμότητας. Ποια θα είναι λοιπόν τα χαρακτηριστικά αυτών των έργων, ποια θα είναι η διάρκεια τους. Τέτοια στοιχεία πρέπει να δούμε. Το Ταμείο θα πρέπει να, το, να λειτουργεί βάσει των αναγκών. ναι, ίσως ε, η Ρουμανία να μην μπορεί να συμβάλλει ε, σε βαθμό 15 εκατομμυρίων στο Ταμείο. Παρ' όλα αυτά είμαι πεπισμένος ότι χρειαζόμαστε στήριξη μέσω αυτού του ε, έργου σχεδίου επενδύσεων. Η Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να συμμετάσχει στην Επιτροπή Επιλογής των Έργων. Τα έργα αυτά θα πρέπει πραγματικά ε, να συμβάλλουν στη γεφύρωση του χάσματο μεταξύ Δύση και ανατολή. Ευχαριστώ. Η κυρία Γιασλουβιέκα ε, είχε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και εγώ ήθελα να συμμετάσχω σε αυτή τη συζήτηση, γιατί όπως πολλοί από εσάς και εγώ συμμερίζομαι αυτές τις ε, αμφιβολίες. Να προσθέσω ακόμα ένα στοιχείο στο χασμό που είναι το κύριο που αφορά την εφαρμογή ε, του προγράμματος και του Ταμείου. Γιατί πολλοί λένε ότι είναι μεγάλα πανευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας, καινοτομίας και του καθεξής. Και λέμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε επενδυτικό κεφάλαιο που έχει που λιμνάζει αυτή τη στιγμή, που ε, ε, μένει παγωμένο. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να δούμε υπάρχει αρκετά μεγάλο δυναμικό ούτω ώστε να συμβάλλουν αυτές οι μικροσές επιχειρήσεις σε τέτοια μεγάλα σχέδια, μεγάλα έργα. Είναι οι μικροσές επιχειρήσεις ικανές γιατί τα περισσότερα κεφάλαια είναι παγωμένα κάπου. Νομίζω ότι είναι δικαιολογημένος αυτός ο προβληματισμός. Αν δούμε μικρές επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη, ίσως να μην είναι έτοιμε για ένα τόσο φιλόδοξο εγχείρημα. Αυτό το σχέδιο επενδύσεων είναι πολύ καλό, αλλά πολύ δύσκολο και συμφωνώ εδώ με ε, τον συνάδελφο από τη Σλοβενία που είπε ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την ε, επιτυχή έκβαση αυτών των επενδύσεων. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Εθνικά Κοινοβούλια, κράτη-μέλη και ούτω καθεξής. Όλοι έχουμε ένα μερίδιο ευθύνη. Αν θέλουμε λοιπόν να αποφύγουμε αυτή την κατάσταση που περιέγραψε προηγουμένω ε, ο συνάδελφο από τη Λιθουανία με τη μετανάστευση των εργαζομένων, και εμεί στην Πολωνία έχουμε ένα παράδειγμα. Νομίζω ότι για να αποφύγουμε κάτι τέτοιο πρέπει να προετοιμάσουμε ήδη από τώρα τι μικροπιστέ επιχειρήσεις ούτως ώστε να δείξουν ενδιαφέρον για την απασχόληση των νέων. Να δίνουμε, να παρέχουμε κάποιο είδου συμβουλευτική, οδηγίε. Αναφερθήκαμε προηγουμένως στις ε, συμπράξει δημοσίου ιδιωτικού τομέα. Νομίζω ο συνάδελφο από τη Λετωνία το ανέφερε. Όμως, ας εξετάσουμε και το εθνικό μας δίκαιο είναι καλοί νόμοι σε εθνικό επίπεδο που μπορούν να στηρίξουν και ε, να ενισχύσουν τις συμπράξεις δημόσιου του δικοτομέα. Εάν όχι, ίσως έχει έρθει η ώρα να διορθώσουμε και το εθνικό μας δίκαιο, να έχουμε ένα ευρύ φάσμα μέσων, ούτω ώστε οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πραγματικά να είναι σε θέση να συμμετάσχουν και αυτό το, και αυτό το στοιχείο της μόχλευσης να μπορέσει να λειτουργήσει. Μετά, από την Πολωνία ένα συνάδελφο. αλλά και ένας ευρωβουλευτής ε, ανέφερε τη μεταφορά των πόρων. Δεν πρόκειται για μεταφορά πόρων. Πρόκειται για, αυτά τα παλιά ε, project που έχουν ήδη ξεκινήσει θα εφαρμοστούν, αλλά θα έχουμε μεγαλύτερη ιδιωτική επένδυση. Σας ευχαριστώ όλους, λέει Πρόεδρος, για τις ε, παρεμβάσεις σας. Βλέπω ότι υπάρχει συνένεση ως προς ότι θα είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, ότι είναι ρηψοκίνδυνο, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα πετύχουμε και ότι όλα μπορούν να πάνε στραβά. Ταυτόχρονα όμως μπορώ να πω ότι μας ενώνει ακριβώς αυτός ο στόχος εδώ στο Κοινοβούλιο αλλά και τα εθνικά κοινοβούλια, ότι είναι μια ανακούφιση, ακόμα κι αν δεν το δούμε στις πατρίδες μας, θα το ακούσουμε εδώ και στα εθνικά μας κοινοβούλια. Δεν συζητούμε μόνο περικοπές και την κατάρριξη της ελπίδα. Μιλάμε και για τις επενδύσεις και το μέλλον. Από κάπου θα πρέπει να ξεκινήσουμε. Αυτό κάναμε λοιπόν, αυτό ξεκινήσαμε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Γιατί δεν είναι μόνο η θέση εργασία ή η νεολαία. Είναι το μέλλον μας, είναι η δημοκρατία. Θα σας ευχαριστώ λοιπόν όλους για τα λόγια σας, για τι ελπίδε σας, αλλά και για την κριτική που εκφράσατε γιατί βεβαίως είμαστε ρεαλιστές. Είμαστε ρεαλιστές, αλλά και με όραμα για το μέλλον. Σας ευχαριστώ όλους.